Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα σας παρακαλέσω να καθίσετε, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι είχαν αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα, κέρδισε τις εκλογές και είστε εδώ. Δεύτερον, συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής, γιατί πρέπει να σας ε, διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ ευχάριστο να είναι κανείς ε, μέλος αυτής της Επιτροπής. Εγώ το λέω από προσωπική πείρα. Και δεν είναι μόνο χαρά, αλλά και τιμή, διότι διατέλεσα πρόεδρος επιτροπής αυτής. Και σήμερα προεδρεύω έστω και προσωρινά και αυτό είναι επίσης μεγάλη τιμή για μένα. Βρίσκεστε σε μια καταπληκτική επιτροπή που έχει πολλές αρμοδιότητες και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Διότι σχεδόν το σύνολο της πραγματικής οικονομίας, οι μεταφορές, βέβαια είναι χαρτοφυλάκιο μιας άλλης επιτροπής, αλλά και μεταφορές εξαρτώνται με θέμα ενέργειας κτλ. Και πλην της Γεωργίας όλες οι άλλες νευραλγικές, νευραλγικοί τομείς εκπροσωπούνται στη δική μας την Επιτροπή. Βλέπω πεπειραμένους συναδέλφους μεταξύ ημών. Συγχαρητήρια να ξεκινήσουμε τη σκληρή μας δουλειά μετά και τις διακοπές. Πρέπει να σας πω ότι εμείς καταφέραμε πριν τις εκλογές να ολοκληρώσουμε με όλα τα νομοθετήματα που σχετίζονταν με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο επιτεύγμα και δεν μπορεί να υπερηφανευτεί για κάτι τέτοιο καμία άλλη από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πριν από τις εκλογές. Ήμασταν οι μόνοι που είχαμε ολοκληρώσει. Ολοκληρώσαμε επίση και τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, το σύνολο των διαπραγματεύσεων που ήταν δική μα αρμοδιότητα. Όλα αυτά πριν τι εκλογές. Και τώρα επανερχόμαστε με σκληρή δουλειά σε πολλού τομείς αρμοδιοτήτων εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα εν γέννη. Λοιπόν, θα τα πω βήμα-βήμα. Είναι μια επίσημη συνεδρίαση αυτή για να βρω τα σωστά χαρτιά. Πρώτα απ' όλα, κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Προφανές αυτό. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά. Θέλω να σας υπενθυμίσω ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής συνεδρίασης. Είναι η συγκρότηση της ομάδας σε, της Επιτροπής σε Σώμα με πρώτο την συγκρότηση του Πρόεδρου, εκλογή Προέδρου και έπειτα ε, εκλογή των Αντιπροέδρων Δυνάμει του άρθρου 213 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι γνωστή η σειρά. Πρώτα εκλέγεται ο πρόεδρος και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου, όμως σε περίπτωση αντικατάστασης, όταν δηλαδή εκπροσωπείται ένας τακτικός ε, βουλευτής από έναν απληρωτή, έχω και τη λίστα εδώ έχουμε το Σον Κέλλη που αντικαθίσταται από τον Ατμαρκάρα, Άλντο Πατριτσέλο που αντικαθίσταται από τον Μασιμιλιάνο Σαλίνη, Αντζέλικα Νίμπλερ αντικαθίσταται από την Ιζαμπέλ Βιζελίμα, Σάρα Σκάιτε Ντίλα από τον Τόμας Τομπέ, η Τερέζα Γκρίφιν από τον Κλοντ Μωράης, Σαν Κόφι αντικαθίσταται από τον Μπρόνις Ροπέ. Τζέφρεϊ Βον Όρντεν. Τζέφρι Φαν Όρντεν. Κροσωπείται από την Λεσπιέτα Κρούκα. Άντρου Ιγκλαντκέρ από τον Ρόλαντ και Τζον Ντέιβιτ Έντουαρτ Τένταντ από τον Αλεξάνδρο Ισλι Φίλιπς. Αυτές είναι οι αντικαταστάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να ψηφίσουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο νομίζω. Δεν ξέρω αν οι πολιτικές ομάδες θέλουν να πούν κάτι. Αν θέλουν να προσθέσουν ή να αλλάξουν κάτι πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές, πριν την κάθε εκλογή. Είναι δυνατόν αλλά πρέπει να μας το πείτε εκ των προτέρων. για να είναι έγκυρη η συνεδρίασή μας. Όταν υπέγραφα, ήμασταν καμιά τριανταριά που είχαμε υπογράψει. Για να έχουμε απαρτία πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 18, άρα είμαστε κατοχυρωμένοι από αυτή την πλευρά. Ένα τέταρτο δηλαδή των τακτικών μελών είναι αρκετό για να έχουμε απαρτία και να προχωρήσουμε στις εκλογές. Λοιπόν, ορισμός Προέδρου. Υποψηφιότητες. είτε πολιτική ομάδα είτε από το 20 των μελών που συγκροτούν την Επιτροπή. Τέσσερα δηλαδή μέλη, τέσσερις βουλευτές αρκούν για να καταθέσουν μια υποψηφιότητα. Και τώρα παρακαλώ να ακούσουμε τις υποψηφιότητες. Έχετε το λόγο. Εσείς παρακαλώ. Κύριος Κρίσταν Χέλερ. την κυρία Βαλεάν έχω την τιμή να προτείνω. Κυρία Αντίνα Βαλεάν λοιπόν είναι η πρόταση. Ε, Αντίνα, δέχεστε να είστε υποψηφία. Ναι, δέχομαι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. έχουμε την αποδοχή της ε, υποψηφίου. Ερωτώ αν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Δεν βλέπω να θέλει να υποβάλει κάποιος άλλη υποψηφιότητα. Έχουμε λοιπόν μία υποψήφια για μία θέση. Πώς θέλετε να ψηφίσουμε, με μυστική ψηφοφορία. Μα τα βλέπω μπροστά μου και τα διαβάζω γι' αυτό, τι να κάνω. Αν 15 βουλευτές ζητήσουν μυστική ψηφοφορία μπορεί να γίνει. Ουδής όμως το επιθυμεί. Σας ευχαριστώ. Τέλεια. Άρα, ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες. Η δυνατότητα εκλογής διαβοής. So, it means... Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ, ήταν καταπληκτικά αυτά τα χρόνια και σας τα λέω ανοιχτά και με κάθε ειλικρίνεια ότι εγώ εδώ ε, σταματώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Αντίνα. Είμαι βέβαιος, Αντίνα, ότι θα είστε μια εξαιρετική πρόεδρος της Επιτροπής Ήτρε. Είχαμε τον Τζάιλς Τσίτσεστερ άντρα. Έπειτα την Αγγέλικα Νίμπλερ, δεν είναι τώρα εδώ. Μετά την Αγγέλικα Ρόμπερτ Ρόιλ. Μετά μια Ιταλίδα βουλευτής. Εγώ, προτελευταίος και τώρα Ρουμάνα, πρόεδρος. Δεν υπάρχει ε, πιο εξαιρετικό παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ των δύο φίλων. Σου εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία αγαπητή Αντίνα και σε καλό να έρθεις ε, στο βήμα για να προεδρεύσεις. Hello everyone. Γεια Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε με την ψήφο σας. Και θα ήθελα όλοι μαζί να καταχειροκροτήσουμε τον Γιέζι Μπούζεκ για τη στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία. Ήταν ένας καταπληκτικός πρόεδρος στην Επιτροπή Ήτρε. Σε ευχαριστούμε θερμότατα, Γιέζι. I'm looking forward to... Ανυπομονώ να συνεργαστούμε όλοι μας εδώ στην Επιτροπή, που είναι πραγματικά συναρπαστική. Και είμαι βεβαία ότι θα έχουμε λόγο και θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της ε, μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής. Γιατί όλοι θα έχουμε ρόλο στην Επιτροπή και ελπίζω να μείνουμε όλοι ικανοποιημένοι. Είμαι βέβαια, μάλλον ευελπίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα και ας μας ευχηθούμε καλή τύχη και καλή επιτυχία στη νέα κοινοβουλευτική θητεία. Επαναρχόμαστε τώρα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίας. Επόμενο μας βήμα είναι η εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής. Έχουμε τέσσερις αντιπροέδρους. Θα εκλέξουμε ξεχωριστά το κάθε αντιπρόεδρο. Περιμένω τώρα τις υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Αν υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα, θα δούμε αν πρέπει να ψηφίσουμε μυστικά ή διαβοή. Αν έχουμε περισσότερου από ανεψηφίου, τότε θα γίνει αναγκαστικά μυστική ψηφοφορία. Αυτό ισχύει. Για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου στην Επιτροπή, ποιο θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα. Το ECR προτείνει τον καθηγητή Κράσινο για πρώτο αντιπρόεδρο. Μάλιστα, κύριε Κρασνοντεύσκη, αυτή είναι η πρόταση του ΕΣΥΑΡ να ε, ε, είστε εσείς υποψήφιος. Άλλη πρόταση υπάρχει για άλλο πρώτο αντιπρόεδρο. Όχι, οπότε να ρωτήσω τον κύριο Κρασνοντέμσκι αν δέχεται την υποψηφιότητα. Μάλιστα, δέχομαι. Ωραία. Ερωτώ την Ομίγυρη, θέλετε μυστική ψηφοφορία ή μπορούμε διαβοή να εκλέξουμε τον κύριο Κρασνοντέμσκι. Ε, για να ζητήσετε μυστική ψηφοφορία θα πρέπει να έχετε 15 ευρωβουλευτές που πρέπει να σηκωθούν και να εκδηλώσουν αυτή την επιθυμία. Σηκωθείτε όσοι θέλετε μυστική ψηφοφορία για να μπορέσουμε να καταμετρήσουμε. 15 χρειάζονται για να γίνει μυστική ψηφοφορία. Δεν αρκεί ο ένας. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρ. Οπότε, διαβοής εκλέγουμε τον κύριο Κρασνοδέμσκι, πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Εξελέγει ο κύριος Κρασνοδέμσκι, οπότε θα ήθελα να τον καλέσω να καθίσει δίπλα μου. Περνάμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες. Η κυρία Ντομπάιωβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και συγχαρητήρια. Και εγώ ως ε, συντονίστρια του Renew Europe ε, αδειμονώ να συνεργαστούμε. Προτείνω το κύριο Μόρτεν Χαλβεκ Πέτερσον ε, για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου γιατί έχει τεράστια πείρα στην Επιτροπή Ήτρε. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι η πρόταση του Renew για την ε, δεύτερη αντιπροεδρία του κυρίου Πέτερσεν. Ο κύριος Πέτερσεν συμφωνεί. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε κύριε Πέτερσεν. Θέλετε μυστική ψηφοφορία. Χρειάζονται όμως 15 μέλη για κάτι τέτοιο. Όχι, οπότε διαβοής. Εκλέγεται ο κύριος Μόρτεν Πέτερσεν, δεύτερος αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ήτρε. Ελάτε κι εσείς στο Προεδρείο. Περνάμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Υπάρχουν προτάσεις για υποψηφιότητες. Ο κύριος Ζωχίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια. Καλή θητεία σας εύχομαι. Επικοδομητική. Και θα ήθελα να προτείνω για τρίτο αντιπρόεδρο κάποιον πυρό, μία γυναίκα μάλλον, τη συνάδελφα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, την κυρία Τόγια, που έχει πολύ πλούσια πείρα. Κυρία Τόγια, δέχεστε ε, την υποψηφιότητα. Μάλιστα, τη δέχομαι. Ωραία. Θέλετε μυστική ψηφοφορία, συνάδελφοι, όχι. Οπότε διαβοής εκλέγεται η κυρία Πατρίτσια Τόγια, τρίτη αντιπρόεδρος. Συγχαρητήρια, κυρία Τόγια. Ελάτε και εσείς εδώ στο Προεδρείο. Και τέταρτος και τελευταίος αντιπρόεδρος, Ποιες είναι οι υποψηφιότητες. Εκ μέρου τη ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητα του συναδέλφου Ζωαμέλα, που ήδη έχει μια πενταετή πείρα ω Ευρωβουλευτή. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρόταση για την υποσύμβα της κυρίας Μέλα. Άλλος υπάρχει κάποια αντιπρόταση, ο κύριος Ζωχίνιο. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες προτείνουν εναλλακτικό υποψήφιο για τη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου, τη Λίνα Γκάλβες, που είναι καθηγήτρια, τακτική καθηγήτρια ιστορίας οικονομίας, ε, είναι δημοτική σύμβουλο στην Ανταλουσία και αυτή είναι η δική μας υποψηφιότητα για τη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου. So now we have a second candidate. Ωραία. Τώρα έχουμε και δεύτερο λοιπόν υποψήφιο. Παρακαλώ πρώτα να μου πούν οι δύο υποψήφιες εάν θέλουν ε, να εκλεγούν. Κυρία Μελάν, δέχεται την υποψηφιότητά της. Μάλιστα. Κυρία Σάλβες Μουνιός. Ναι και ευχαριστώ. Καλώς, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να γίνει εδώ ψηφοφορία με τρόπο ηλεκτρονικό. Παρακαλώ λοιπόν να βγάλετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Είναι στα μηχανήματά σας. like to ask the coordinators to have a check uh, in their teams to see Παρακαλώ τους συντονιστές να επαληθεύσουν ε, ότι οι συνάδελφοι της κάθε ομάδας ε, έχουν όλοι τις κάρτες τους, ότι, είναι, λειτουργούν όλα σωστά. Και να μου κάνουν ένα νεύμα αν όλα πάνε καλά οι συντονιστές. Το ΕΛΚ εντάξει, οι σοσιαλιστές. Δεν βλέπω αντιδράσει, επομένω φαντάζομαι ότι όλα πάνε καλά. Θα κάνουμε το εξή. Το πράσινο κουμπί για την κυρία Μελά, το κόκκινο για την κυρία Σάλβες Μούνιος. Και αν θέλετε να δηλώσετε αποχή, λευκό, αλλά δεν προσμετρούνται οι αποχές, για τις πλειοψηφίες που απαιτούνται. Η πλειοψηφία είναι απλή με βάση τα έγκυρα, τις έγκυρες ψήφους. Έγινε σαφές. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πράσινο για την κυρία Μελά. Κόκκινο για την κυρία Κάλβας Μούνιος. Um, did everyone voted? Ψήφισαν όλοι. See any... Okay, then the vote is closed. Πέρας. So we have 69 votes expressed. Ψήφισαν λοιπόν 69, τρεις ήταν οι εποχές και πλειοψηφία επομένως επί 66. Θα χρειάζονταν ως εκ τούτου 33 συν μία ψήφη. Η κυρία Κάλβες Μούνιος κερδίσε εξελέγη και συγχαρητήρια. Uh, dear colleagues, Σας συγχαίρω και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Και πριν κήρυξω το πέρα στη συνεδριάσεως, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως η προσεχή μας ε, συνεδρίαση βλέπετε για τις 23 Ιουλίου στις Βρυξέλλες με φιλανδική προεδρία ήδη. Και αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας περιμένω λοιπόν 23 του μηνός στις Βρυξέλλες. Καλό σας απόγευμα.